τακτική να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να παίξει εκεί σημαντικό ρόλο. Ε, το 2012 ε, μπορεί ε, να είναι κρίσιμο έτος για την Ισλανδία διότι η Ισλανδία επιθυμεί να ανοίξει το συντομότερο δυνατόν όλα τα κεφάλαια υποδιαπραγμάτευση και κάποια στιγμή να κλείσουν και αυτά εν το χρόνο. Κυρία Πρόεδρε, καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή, λέει ο κύριος για την έκθεσή του εγώ ήμουν μέλος ε, της αντιπροσωπείας που επισκέφθηκε την Ισλανδία και δεν είχα ξαναπάει, δεν περίμενα να δω τίποτα άλλο παρά μόνο κάποια βράχια και ερημιά, αλλά τελικά πράγματι είναι ένα πολύ ενδιαφέρον μέρος ε, και εκεί συναντήσαμε και πολύ ενδιαφέροντες πολιτικούς. Κατόπιν τούτου θα ήθελα να φερθώ σε ένα-δύο σημεία, αν μου επιτρέπετε. Εγώ δεν έχω διαφορετική άποψη από την έκθεση του εισηγητή. Εντάξει, κάποιες αποκλίνουσες αποχρώσεις, αλλά να πω το εξή. Συναντηθήκαμε, παραδείγματος χάρη, με τον Υπουργό Αλίας, ο οποίος, ε, κατά την άποψή μου, είναι άκαμπτος, ε, είναι ο πιο άκαμπτος σταλινιστής που έχω συναντήσει ποτέ σε δημοκρατική χώρα. Είπε λοιπόν αυτός ότι για να μπει χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να περάσει πάνω από τα πτώμα του. Και το είπανε και άλλοι. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να πούμε ότι στην Ισλανδία υπάρχει διάσταση απόψεων. Ε, μας είπαν ότι στην τελευταία ε, κλείνει λιγάκι το χάσμα, 50% είναι υπέρ, 50% ε, κατά, ενώ παλιά η ε, κατά ήταν περίπου στο 75%. Ένα πράγμα λοιπόν που με εντυπωσίασε και το είπα αυτό σε κάποιο άτυπο εκεί δείπνο που είχαμε, το είπα στους συντηρητικούς επικεφαλής κομμάτων. Από ό,τι φαίνεται ε, δεν έχουν καν αποφασίσει κατά πόσο να τα υποβάλουν επίσημα την αίτηση, πόσο μάλλον να ενταχθούν. Αυτό που με εντυπωσίασε είναι ότι δεν έχουν καταλήξει ακόμα εκεί. Γιατί, μάλλον, υποτίθεται ε, επίσημα έχουν ε, υποβάλει την έτσι, αλλά δεν έχουν καταλήξει αν θέλουν ή όχι. Τώρα, το να ε, διοργανώσουν δημοψήφισμα, αυτό θα σημαίνει ότι πρέπει να περιμένουν το αποτελέσμα, το, το αποτέλεσμα των ε, διαπραγματεύσεων, μετά να κάνουν ε, την αίτηση συνέχεια, ε, ξανά διοψηφίσμα. Τέλο υπάρχει μια πολύ μεγάλη σύγχυση και δεν έχω καταλάβει ακριβώ τι θέλουν οι άνθρωποι αυτοί. Και όπω είπε και ο εισηγητή, το κύριο ε, κυβερνών κόμμα τάσεται αναπιφύλακτα υπέρ τη ένταξη, ενώ ε, το συνεργαζόμενο κόμμα είναι κατηγορηματικά κατά τη ένταξη. Και όταν το θέμα τέθηκε στο Κοινοβούλιο, η κυβέρνηση συμμαχίας πήρε την υπερψήφιση μόνο με μία ψήφο υπέρ και έγινε αυτό κυρίως για να διατηρηθεί η κυβέρνηση. Υπάρχει λοιπόν έντονη διάσταση απόψεων για το τι επιθυμούν να κάνουν. Ένας από τους ε, βουλευτές ε, που ασχολείται με τα οικονομικά είπε ότι θέλει σαφώς να μπει στο ευρώ. Το είπε τότε, δεν ξέρω αν το έλεγε σήμερα, τότε ήταν σαφώς υπέρ του ευρώ και υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό από μόνο του λέει πολλά. Έτσι λοιπόν λοιπόν ο εισηγητής ε, σωστά επισημαίνει και τα προβλήματα με την Αλία και τη Γεωργία. Ε, στην ε, Γεωργία υπάρχει μια μετακίνηση, αλλά δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε τελικά να βρούμε ένα μόντους βιβέντη για την Αλία. Γιατί η Αλία είναι το α και το ω της οικονομίας, πόσο μάλλον του πολιτισμού της Ισλανδίας. Και το να τους ε, ζητάμε αυτά που τους ζητάμε αυτή τη στιγμή, αυτό είναι απαράδεκτο. Έτσι λοιπόν οι διαπραγματεύσεις ε, ε, θα είναι να δούνε και λαβίν και όπως μας είπε και ο συνάδελφος Στίβενσον υπάρχει και το πρόβλημα το μακροοικονομικό. Πρέπει και αυτό να το λύσουμε. Ο κύριος Στίβενσον εκπροσωπεί βέβαια τη Σκοτία και έχει από αυτού άκαμπτες απόψεις. Ε, έτσι λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, σε γενικέ γραμμέ ε, συμφωνώ με τον εισηγητή. Υπάρχουν μόνο δύο άλλα θέματα που θέλω και αυτά να δείξω και είναι καθοριστική σημασία. Η άμεση επιστροφή του χρέους πρόκειτο να λάβει χώρα. Αυτό πιστεύαμε. Και αυτό μου είπανε και κάποιοι εκπρόσωποι ε, της ε, τοπικής οδίκης στη Βρετανία. Βέβαια αυτοί πληρώθηκαν από την κυβέρνηση αλλά μου είπαν ότι η Ισλανδία ήδη πληρώνει κάποια χρήματα στην ε, Μεγάλη Βρετανία. Αυτό που ενδιαφέρει είναι να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα στην Αρκτική. Η Ισλανδία ως μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έπαιζε σημαντικό ρόλο στις σχέσεις στο θέμα της Αρκτικής. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό είναι από τα καθοριστικά θέματα το οποίο πρέπει να προβάλλουμε στις διαπραγματεύσεις με την Ισλανδία. Έτσι λοιπόν και πάλι συγχαρητήρια στον εισηγητή. Δεν υπάρχει πρόβλημα με την ουσία της έκθεσης και το έχουμε καλή επιτυχία. Η κυρία Σαρτζεντίνη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ήμουνα με τον εισηγητή του Πρέντα στο ταξίδι. Πρώτη φορά πήγα στην Ισλανδία και έμαθα πολλά από την επίσκεψη αυτή. Αυτό όμως που με έκανε κυρίως εντύπωση είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή, το Κοινοβούλιο θέλουν πάρα πολύ την Ισλανδία να ενταχθεί Είχαμε τη συζήτηση πριν για την Τουρκία, έτσι, μην το ξεχνάμε. Παρ' όλα αυτά τα πράγματα είναι κάπως περίπλοκα. Η Ισλανδία ως χώρα έχει πληγεί πάρα πολύ από την οικονομική κρίση και αποτελεί μέρος μια ομάδα χωρών που επίσης υποφέρουν από την οικονομική κρίση. Εμάς ε, μας ε, έκανε πολύ εντύπωση. Γι' αυτό και τους φαίνεται το ευρώ που έχουμε εμείς εδώ σαν κάτι ελκυστικό. Υπάρχουν αλλαγές στην ε, ε, κοινή γνώμη πάντως για το θέμα της ένταξης της Ισλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει το σημείο 9 στο ψήφισμα αυτό, το οποίο κάτι αλλάζει. Αν θέλουμε εμείς να βοηθήσουμε την κατάσταση στην Ισλανδία. Εμείς πρέπει να πούμε ότι σημειώνουμε την κατάσταση εκεί. Η διαφορά πάντως είναι ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να προχωρήσει και να λειτουργήσει και κινδυνεύουν να σταματήσουν οι διαπραγματεύσεις. Η αντιπολίτευση στην Ισλανδία είναι εκείνη που θέλει να σταματήσουν οι διαπραγματεύσεις. Εμείς πρέπει να δείξουμε κάθε σεβασμό στην κυβέρνηση της ε, Ισλανδίας ώστε να υπάρχει κάποια ισορροπία για το θέμα της ε, ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κρίμα που υπάρχει πάντα το πρόβλημα με το σκουμπρί. η κυβέρνηση πρέπει να μπορέσει να διαχειριστεί καλύτερα τα δικά της τα ύδατα όσον αφορά την αλίευση. Για μας τους πράσινους επίσης το θέμα ε, της φάλαινας είναι κάτι που μας απασχολεί πολύ. Και μου έκανε φοβερή εντύπωση όταν μου φέραν σε ένα πιάτο κρέας φάλαινας να φάω. Για μας καταλαβαίνετε ότι είναι πρόβλημα. Και για να μιλήσω και για κάτι θετικό, πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να υποφεληθεί όσον αφορά την ενέργεια, διότι έχει ε, μονάδες υδροελεκτρικής ενέργειας στη Ισλανδία και από αυτό μπορεί να υποφεληθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Πουντζέρη. Ναι, από ο κύριος δεν είναι εδώ σήμερα. Α, η υποκυρία Ζολή δεν είναι εδώ σήμερα, συγγνώμη όπως ε, σας είπα, ε, αντικαθέτω τον κύριο Σασόλη. Και θα ήθελα να πω ότι η εισήγηση του κυρίου Πρέντα είναι πάρα πολύ καλή και εξετάζει όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την ε, Ισλανδία. Το κείμενο του ψηφίσματος εμεί το αντιμετωπίζουμε θετικά και πρέπει πράγματι να υπογραμμίσουμε ότι η Ισλανδία έχει σημειώσει πρόοδο, κυρίως όσον αφορά στην ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας. Επίσης είναι πολύ θετικό το ότι έχουν ανοίξει έξι ε, κεφάλαια ε, και έχουν κλείσει προσωρινά τέσσερα. Αυτό δείχνει δηλαδή ότι η χώρα επιθυμεί να προχωρήσει σε αυτό το δρόμο της ένταξης. Υπάρχουν αυτά τα θετικά, όμως υπάρχουν και κάποιες σκιές που πρέπει να διαλευκανθούν. Ε, υπάρχουν προβλήματα που ετέθησαν ήδη επιτάπητος. Κυρίως όσον αφορά στο θέμα ΆΙΣΕΒ e Αυτό πρέπει να λυθεί. Η Ισλανδία είναι α, το, η οποία πρέπει να προχωρήσει το θέμα αυτό σχετικά με την Ice Save. Επίσης, ε, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ε, η πολιτική αλίας βρίσκεται σε φάση μεταρρύθμισης. Ε, έτσι θα πρέπει να επιτευχθεί μια συμφωνία που να ικανοποιεί και τις δύο χώρες πρέπει πράγματι να ε, γίνεται σεβαστή εκμετάλλευση των αληφτικών πόρων και η διατήρηση των θέσεων στον τομέα της αλίας. Ε, η ε, φαλαινοθυρία αυτό είναι ένα θέμα που επίσης πρέπει να συζητηθεί στο πλαίσιο της μελλοντικής συμφωνίας. Τελειώνοντας, ε, πρέπει να πω ότι σημειώθηκε σημαντική πρόοδος και η πρόοδος αυτή έχει καταδείξει ότι υπάρχει βούληση να συνεχιστούν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Εμείς ε, ως ομάδα των σοσιαλιστών και των δημοκρατών θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε το άνοιγμα των διαφόρων κεφαλαίων, θα συνεργαστούμε με τον εισηγηστή και θα καταθέσουμε κάποιες ε, τροπολογίες οι οποίες όμως θα ακολουθούν τον δρόμο που χαράσει εκείνος ο εισηγητής. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Γκόμες, η Άννα. Euh, euh, Θέλω να χαιρετήσω τον συνάδελφο Πρέντα για την εκθεσή του και νομίζω και εγώ ότι ενισχύει πολύ τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Α, γιατί από ό,τι γνωρίζω εγώ, γιατί δεν ήμουν στην, επίσκεψη, την μία της επίσκεψης, Γνωρίζω όμως την Ισλανδία και εκτιμώ ιδιαίτερα, θαυμάζω τη χώρα αυτή και τον λαό της. γιατί έχει πολύ ισχυρή δημοκρατία, ριζωμένη δημοκρατία και σέβεται πολύ τα ανθρώπινα δικαιώματα και έζησε και την κρίση την, στην οποία, από την οποία βγήκε επιτυχώς. Με πλήρη σεβασμό της των δημοκρατικών διαδικασιών. Και άλλοι είπαν ότι η εμπειρία της Ισλανδίας για τις ανανεώσιμες, ιδίως τη γεωθερμική ενέργεια, είναι επίσης κάτι ιδιαίτερα ωφέλιμο θα είναι για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κλιματολογικές αλλαγές στην Αρκτική είναι επίσης κάτι που το γνωρίζουν οι Ισλανδοί. Ξέρουμε ότι οι Πορτογάλοι καταναλώνουν ιδιαίτερα μεγάλες ποσότητες βακαλάου και αυτός προέρχεται κυρίως από την Ισλανδία. Θα έπρεπε ίσως να αναμορφώσουμε όλη μας την αλληλευτική πολιτική για να βρούμε μια λύση που να ικανοποιεί και τις θεμητές ανησυχίες των Ισλανδών. Υποστηρίζω λοιπόν τα συμπεράσματα του συναδέλφου Πρέντα. Ευχαριστούμε ο κύριος Ντάρτμουντ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ έχω κάποιες παρατηρήσεις να κάνω. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πω, ίσως να μην ακούστηκε καλά προηγουμένως, αλλά ο συνάδελφος ε, που είναι επίσης αναπληρωτής ε, μοιάζει να έκανε την παρατήρηση ότι η Ισλανδία έχει να μάθει από την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την βιώσιμη αλία. Εγώ αυτό άκουσα, αλλά πρέπει να πω ότι μπορεί κανείς ε, να μάθει κάτι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η έννοια, κυρίως ε, για την Αλία, όπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα νεκρά ψάρια ξαναρίχνονται στη θάλασσα, καταλαβαίνετε αυτό ε, είναι ηρωνία. Η δική μας η Αλία καταστράφηκε με την ε, ένταξη ή λόγω του γεγονότος είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Άτκινς ε, ήταν ε, ιδιαίτερα αρνητικός όσον αφορά τις απόψεις του Υπουργού Αλίας στην Ισλανδία. Τον χαρακτήρισε μάλιστα σταλινιστή. Αλλά εγώ πρέπει να σας πω ότι αν είναι κανείς υπουργό Αλίας της Ισλανδίας, το ελάχιστο που μπορεί να κάνει, και εδώ παρεπιπτόντως η Ισλανδία είναι πολύ πιο ανεξάρτητη για την Αλία από οποιαδήποτε άλλη οικονομία του κόσμου, είναι λοιπόν ε, απόλυτα σωστό να είναι κανείς τουλάχιστον επικριτικός κυρίως ως προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το να τον λέει κανείς σταλινιστή απλά επειδή διαφώνησε με τον Ρόμπερτ Άτκινς, ε, εντάξει τι να πω. Να υπενθυμίσω επίσης τον κύριο Άτκινς ότι η Ισλανδία έχει κοινοβούλιο για πάνω από χίλια χρόνια. Κάποιος λοιπόν τώρα που έρχεται από ένα κοινοβούλιο που υπάρχει για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, το να λέει σε έναν άλλον που διαφωνεί μαζί του ε, ότι είναι σταλινιστής, δεν θα πω τίποτα άλλο θα πω κάτι άλλο που είναι πολύ πιο σημαντικό κατά την άποψή μου. Σχετικά με τη διεύνηση, η Ισλανδία είναι υποψήφια χώρα. Ε, το γεγονός είναι ότι οι πλούσιες χώρες όπως η Ελβετία και η Νορβηγία δεν θέλουν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οι φτωχές όπως η Κροατία, το Κοσφοπέδιο, υποθέτω και η Σερβία, το Μαυροβούν. Αυτές φλέγονται, θέλουν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την Ισλανδία έχουμε λοιπόν ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα που στηρίζει αυτήν την την παραδοχή τη δική μου. Η Ισλανδία ήταν μια πλούσια χώρα και έτσι θεωρεί τον εαυτό τη. Όταν ήταν πλούσια χώρα, όπως είπε ο Σερ Ρόμπερτ περίπου 80% των πολιτών ήταν κατά της ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μετά ήρθε η χρηματοψηφιακή κρίση, η οποία χτύπησε την Ισλανδία χειρότερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Και κάτω από αυτές τις ε, καινούργιες ε, συνθήκες όπου η Ισλανδία πλέον θεωρεί ότι είναι φτωχή χώρα άλλαξε άποψη και βέβαια ε, υπάρχουν διστάμενες απόψεις από αυτού. Τώρα η Ισλανδία λόγω της εφευρετικότητας του λαού της που αναφέρθηκε προηγουμένως και βεβαίως και λόγω ε, του ότι η αλία της είναι ιερή, λόγω αυτών η, Ισλανδία ανέκαμψε και μάλιστα επιστρέφει και χρήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο, κάτι που είναι σχεδόν ασυνήθιστο με έννοιες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα λοιπόν θεωρεί η Ισλανδία ότι είναι σε καλύτερη οικονομική θέση. Και τι σημαίνει αυτό, ο αριθμός, το ποσοστό αυτών που είναι υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης μειώνεται. Έχουμε φτάσει στο 50-50. Ως λοιπόν η Ισλανδία θα συνεχίσει να προοδεύει και είναι όλο και πιο επιμερούσα, όλο και περισσότεροι άνθρωποι θα είναι κατά της ένταξης. Εγώ λέω λοιπόν στους Ισλανδούς, αν θέλετε να μπείτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μην το κάνετε. Θα σας καταστρέψουν την αλία, θα γίνετε καθαρό συνεισφορέας, θα πληρώνετε για να στηρίζετε χώρες όπως είναι το Κοσμοπέδιο, να μην το κάνετε σας λέω εγώ. Να γνωρίσετε τους ε, πολιτικούς σας και κυρίως να γνωρίτε τους ε, επισκέπτες πολιτικούς που έρχονται σε και όσοι διαφωνούν τους αποκαλούν σταλινιστές. Merci. Ευχαριστούμε κύριε Ντάρτμοντ. Βλέπετε ότι σας αφήνουμε να εκφραστείτε ελεύθερα όταν σέβεστε το χρόνο σας. Η κυρία Σαργεντίνη θα σας απαντήσει. Ναι, στα αγγλικά όμως, γιατί είδα ότι όταν μιλάω Ολλανδικά δεν με καταλαμβάνετε. Λοιπόν, για τη βιώσιμη αλληλεία δεν εννοούσα ότι η Ισλανδία μπορεί να πάρει μαθήματα από εμά, αλλά το ανιντίθετο. Ο κύριος Βίγκενιν. Ευχαριστώ. Ήθελα να αλλάξουμε ύφος και να πω το εξής. Συχνά όταν μιλάμε για διεύρυνση, μιλάμε για, εννοούμε τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και ξεχνάμε ότι και η Ισλανδία είναι χώρα που ήδη διαπραγματεύεται πιθανή ένταξη. Και προσπαθούμε στις σχέσεις μας με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων να έχουμε ένα συνεχή πολιτικό διάλογο και οι συνάδελφοί μας από την Ισλανδία παρεξηγούνται ότι έχουν την εντύπωση ότι δεν μας ενδιαφέρει η Ισλανδία. Με την Ισλανδία δεν υπάρχουν και πολλά προβλήματα βέβαια, αλλά πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να αυξήσουμε τον διάλογο μας, την παρουσία μας εκεί, και οι πολιτικές ομάδες του Κοινοβουλίου μας να αυξήσουν τις σχέσεις τους, να γνωρίσουν τι θέλει και τι δεν θέλει η Ισλανδία, να υπάρχει ένας καλύτερος διάλογος. Βέβαια τελικά ο λαός της Ισλανδίας θα αποφασίσει αν θέλει να ενταχθεί στην Ένωση ή όχι. Αλλά η σχέση που ανέφερε ο κύριος Ντάρτμοντ ότι μια χώρα όταν είχε δυσκολίες ήθελε να μπει και όταν έπαψαν οι δυσκολίες δεν θέλει πια. Είναι κάτι απλοϊκό σαν αντίληψη της ένταξης. Το θέμα δεν είναι μόνο οικονομικό. Πρέπει αυτό να το ξεκαθαρίσουμε στους πολίτες της Ισλανδίας από τώρα. Αλλά είναι θέμα, θέμα αλληλεγγύης, κοινών στόχων, και δεσμεύσεων και αν παρουσιάσουμε την Ένωση μόνο σαν έναν κατανομέα χρημάτων, ε, τότε φυσικά θα ενδιαφέρονται λιγότερο οι πλουσιότερες χώρες να μπουν σε τέτοια Ένωση. Να εξηγήσουμε λοιπόν τι ακριβώς είναι η Ένωση και να μην τα λέμε απλοϊκά. Ευχαριστούμε τώρα ο εισηγητής ο κύριος Πρέντας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για όσα είπαν και τα σχόλιά τους. Δεν τέθηκε κανένα ερώτημα ή απορία, αλλά το θέμα για την αλληλεία δεν θέλω να αναφερθώ σε ενδοβρετανικές συζητήσεις ο Άτκινς Ντάρτμουθ. Δεν είναι ο ρόλος μου αυτός. Απλώς θέλω να σας παραπέμψω στα στοιχεία μιας πρόσφατης δημοσκόπησης στην Ισλανδία που δείχνουν ότι δύο τρίτα θέλουν να φύγει ο Υπουργός Αλληλείας διότι δεν θεωρούν ανίκανο πλέον να διαχειριστεί το θέμα του. Και προτείνει η Ιρλανδία η αλληλεία να συμπεριληφθεί στο υπου, αρμοδιότητες του Υπουργείου Βιομηχανίας και Τουρισμού. Για αυτά που είπε η κυρία Σαργεντίνη. Τις διαφορές αυτές που υπάρχουν μέσα μεταξύ των υπουργών πρέπει να τις πούμε, να μην τις κρύψουμε. Αλλά δεν νομίζω ότι η έκφραση που χρησιμοποίησα ήταν ιδιαίτερα οξία, ίσα ίσα. Είπα, είναι πολύ ενδιαφέρον πολιτικό φαινόμενο, ιδιαίτερα διότι αν δούμε τι έγινε στις τελευταίες διευρύνσεις. Για τον Σκόμβρο είναι κάτι που μας διαιρεί στη συζήτηση μας με την Ισλανδία και φαντάζομαι ότι δεν θα παίξει ιδιαίτερο ρόλο στις διαπραγματευτικές, στις ενταξιακές όμως διαπραγματεύσεις. Συμφωνώ απόλυτα με την κυρία Σερτζαντίνη πάντως και με τους άλλους που είπαν ότι η Ισλανδία αποτελεί πηγή έμπνευση για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό ναι, και μπορούμε να περιμένουμε πολλά σε αυτό το τομέα. Ευχαριστώ πάντως και τον κύριο Πατζέλη και την κυρία Γκόμες για τις παρατηρήσεις τους σχετικά με το θέμα αυτό της Ισλανδίας και ευχαριστώ και τον κύριο Βιγγένιν που υπενθύμησε ότι η Ισλανδία μπορεί να μην είναι Δυτικά Βαλκάνια είναι όμως πάντα μια υποψήφια χώρα. Είναι μια ειδική περίπτωση λοιπόν. Δεν έχει να κάνει κατά τη γνώμη μου με τη φτώχεια ή τον πλούτο και όσον αφορά την παρατήρησή σας για την στήριξη στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, να ξέρετε ότι η στήριξη αυτή ήταν μεγαλύτερη πριν από την κρίση. Δεν είναι μετά την κρίση που στηρίχθηκε περισσότερο το θέμα της ε, ένταξης. Το θέμα της σταθερότητας του ευρώ καταλαβαίνετε ότι δεν αποτελεί πια ε, επιχείρημα. Δεν είναι οι Ισλανδοί οι οποίοι θα βοηθήσουν να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη στο ευρώ. Άρα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Η στήριξη υπήρχε πριν την κρίση για την ένταξη. Κατά τη διάρκεια της κρίσης είναι αλήθεια ότι οι σοσιαλιστές στην Ισλανδία, οι σοσιαλδημοκράτες επωφελήθηκαν ώστε να συζητηθεί το θέμα στη Βουλή. Πάντως η μείωση της εμπιστοσύνης στην Ευρώπη έχει να κάνει με την αποδυνάμωση του ευρώ. Δεν έχει να κάνει με τη σχέση φτώχειας πλούτου ήθελα να τις κάνω αυτές τις διευκρινήσεις. Τέλη Ιανουαρίου θα ξανασυζητήσουμε. Και σίγουρα θα μας πείτε εσείς κύριε Πρόεδρε πότε ακριβώς. Ευχαριστούμε κύριε Πρεντάλη Πρόεδρος. Ναι. Υπενθυμίζω λοιπόν τις ημερομηνίες. Σήμερα είχαμε την πρώτη ανταλλαγή. Προθεσμία είναι 12 Ιανουαρίου στις 12 το μεσημέρι για την κατάθεση τροπολογιών. 31 Ιανουαρίου θα συζητήσουμε πάνω στις τροπολογίες, θα ψηφίσουμε εδώ στις 6 Φεβρουαρίου και στην Ολομέλεια τον Μάρτιο. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή για την ε, δουλειά του. Και περνάμε στο σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης που είναι η συμμετοχή του Βασιλείου του Μαρόκου στα προγράμματα της Ένωσης είναι ένα σχέδιο σύστασης για ένα πρωτόκολλο στη Συμφωνία Σύνδεσης Ευρωπαϊκή Ένωση Μαρόκου που επιτρέπει στο Βασίλειο του Μαρόκου να συμμετέχει στα κοινοτικά προγράμματα. Το πρωτόκολλο το οποίο τίθεται προς έγκριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βασίζεται στις γενικές αρχές συμμετοχής στα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Μαρόκου. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Νέιτς, η οποία είναι και η συγκήτρια. Παρακαλώ κυρία Νέιτς, είχατε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα, να σας πω κάποιες οργανωτικές λεπτομέρειες. Όταν έφτασα εδώ, οι κύριοι που σέρβιραν καφέ ήταν ε, έξω, είχαν ήδη βγει από την αίθουσα και αρνήθηκαν να ξαναμπούν για να μου σερβίρουν καφέ. Οπότε βγήκα για να πάρω καφέ εγώ έξω. Ίσως θα πρέπει να τους ζητήσουμε να δείχνουν κάπως μεγαλύτερη ευγένεια απέναντι στους ευρωβουλευτές. Εντάξει, δεν λέω ότι είναι σημαντικό, αλλά ήθελα να σας το έχω πει. Έρχομαι τώρα στην νομοθετική αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, υπάλληλοι από τις διάφορες πολιτικές ομάδες, παρακαλώ ησυχία. Ναι, μπορείτε παρακαλώ. Θα ήταν πολύ καλό αν τα πηγαδάκια σας τα κάνατε έξω και όχι μέσα στην αίθουσα. Λοιπόν, μιλάω για την ευρωπαϊκή πολιτική γυτνίασης. ανοίγουν σιγά σιγά κάποια προγράμματα και κάποιοι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ε, χώρες εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πολιτική γετνίαση. Είναι ένα από τα πολλά μέτρα που υιοθετούμε για να στηρίξουμε τον εξυγχρονισμό και την ε, μεταπολίτευση σε γείτονες χώρες μας. Οι στρατηγικοί στόχοι αναφέρονται στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τη γενική προσέγγιση που έχουμε από το 2007 και έχει εγκριθεί στις 5 Μαρτίου 2007 από το Συμβούλιο. 18 Ιουνίου του 2007, βάσει της ανακοίνωσης αυτής και βάσει των συμπερασμάτων, το Συμβούλιο ε, ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις για διάφορες συμφωνίες πλαίσιο με διάφορες γείτονες χώρες, μεταξύ άλλων και το Μαρόκο. Και συμφωνίες αυτές πλαίσιο βασίζονται στις γενικές αρχές συμμετοχής τους στα κοινοτικά προγράμματα. Ένα επιπλέον πρωτόκολλο κατέληξε το 2007 με το Ισραήλ και στη συνέχεια υπογράφηκε τον Απρίλιο του 2008 ένα άλλο τέτοιο πρωτόκολλο και έχουμε και τη συμφωνία με την Ουκρανία που έχει επίσης καταλήξει. Στη συνέχεια αποφασίστηκε να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με το Μαρόκο, οι οποίες κατέληξαν προς ικανοποίηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αποτελούν αντικείμενο νομοθετικής πρότασης της 17ης Μαΐου του 2010 και εγκρίθηκε μετά τροποποίηση δίχως άλλο, από το Συμβούλιο το Σεπτέμβριο που μας πέρασε. Και το Συμβούλιο έχει ήδη δημοσιεύσει μια νομοθετική πρόταση στις 27 Σεπτεμβρίου. Η νομική βάση είναι το άρθρο 217 της συνθήκη της Λισαβόνας, παράγραφος 6, σημείο 1 και παράγραφος 8, δεύτερο εδάφιο. Το πρωτόκολλο επικεντρώνεται στις γενικές αρχές συμμετοχής του Μαρόκου στα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιο συγκεκριμένα σε προγράμματα που έχουν να κάνουν με κατά προτεραιότητα τομείς τόσο για το Μαρόκο όσο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι η ανταγωνιστικότητα και η καινοτομία, τα τελωνία, το Σέζαρ και το Μάρκο Πόλο. Το πρωτόκολλο περιλαμβάνει διάφορες ε, αρχές που έχουν να κάνουν με τη συμμετοχή στα κοινοτικά προγράμματα του Μαρόκου. Και ιδιαίτερα αναφέρονται οι τρόποι, οι ειδικέ προϋποθέσεις που εφαρμόζονται στη συμμετοχή του Μαρόκου σε κάθε ιδιαίτερο πρόγραμμα. Ιδιαίτερα αναφέρεται η οικονομική συμμετοχή, ναι. καθώς και οι διαδικασίες αξιολόγησης που μένει να ε, συμφωνηθούν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δράει εκ μέρου Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μαρόκο. Επίση, προβλέπεται ότι προ το παρόν ισχύουν οι διατάξει του πρωτοκόλου τη ημερομηνία τη υπογραφή. Δεν ξέρω τώρα αν χρειάζεται να σας απαριθμίσω τις διάφορες διατάξεις του πρωτοκόλου αυτού. Το βασικό είναι ότι επιτρέπει στο Μαρόκο να συμμετέχει σε όλα τα σημερινά και μελλοντικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, συνεσφέρει το Μαρόκο οικονομικά στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, βάσει των ειδικών προγραμμάτων στο οποίο συμμετέχει. Οι εκπρόσωποι του Μαρόκου επίσης ε, δικαιούνται ως παρατηρητές να συμμετέχουν για τα σημεία τα οποία τους αφορούν στην Διαχειριστική Επιτροπή που παρακολουθεί τα προγράμματα αυτά οι πρωτοβουλίες από πλευράς του Μαρόκου τίθενται στους ίδιους κανόνες και διαδικασίες ή δυνατόν, όπως και, δηλαδή συμμετέχει με τους ίδιους όρους όπως και οι χώρες μέλη στα προγράμματα αυτά. Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, η οικονομική συνεισφορά και οι διαδικασίες αξιολόγησης καθορίζονται στα πλαίσια μιας συμφωνίας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αρχές του Μαρόκου. Και ότι οι οικονομικοί έλεγχοι θα πρέπει να πραγματοποιούνται και επίσης ότι ισχύει το πρωτόκολλο για την περίοδο κατά την οποία η ε, σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης Μαρόκου εξακολουθεί να ισχύει. Δεν έχει επιπτώσει στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί το Μαρόκο συνεισφέρει οικονομικά στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναλογικά στο επίπεδο δηλαδή που συμμετέχει στα επιστημονικά προγράμματα. Μπορεί όμως να ζητήσει αρρωγή βάσει του κανονισμού που έχει να κάνει με το Ευρωπαϊκό Μέσο Γυτνίασης που ήδη ισχύει. Συνεπώς, η πρόταση που σας υποβάλλω σήμερα, σήμερα. να σημειώσω εδώ ότι ό,τι έχει να κάνει με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες αποτελεί ένα πολύ σημαντικό στοιχείο στις σχέσεις μας, Ευρωπαϊκή Ένωση Μαρόκο δηλαδή, και ότι η συμμετοχή του Μαρόκου σε αυτά τα διάφορα προγράμματα πρέπει να ε, βοηθήσει όλο τον πληθυσμό, όλη την επικράτεια, δηλαδή συμπεριλαμβανομένης και της Δυτικής Σαχάρας. Ξέρω ότι αυτά είναι θέματα που δημιουργούν μεγάλες ανησυχίες όλους τους συναδέλφους και σε μένα την ίδια. Πιστεύω όμως ότι θα έπρεπε αυτό να διευκρινιστεί. Και προτείνω να συμφωνήσουμε με το πρωτόκολλο αυτό Ευρωπαϊκής Ένωσης Μαρόκου. Τώρα επιτρέψτε μου να κάνω και ένα τελευταίο σχόλιο προσωπικό, κυρία Πρόεδρε, σύντομα. Θέλω να υπογραμμίσω Λέγοντα ότι γνωρίζω καλά το Μαρόκο. Πολύ συχνά πηγαίνω, το γνωρίζω καλά. Θέλω λοιπόν να υπογραμμίσω ότι δεν θα πρέπει να τιμωρούμε το Μαρόκο επειδή δεν πέρασε από τις ταραχές που είδαμε βλέπουμε ακόμα στην Αίγυπτο και σε άλλες χώρες της περιοχής. Βλέπετε το Μαρόκο ξεκίνησε τις ε, μεταρρυθμιστικές του διαδικασίες εδώ και πολλά χρόνια. Εφαρμόζοντας αποφάσεις του Μωαμέτ, ε, του Μωαμέτ του Έκτου, θα θυμόσαστε ότι υπήρξε διαφάνεια, συμφιλίωση σε σχέση με ε, την εποχή του Μολύβου, όπως τον λένε, τα παριά χρόνια εκείνα. Ο βασιλιάς πάντως δύο φορές άλλαξε τον νόμο για τις γυναίκες. Υπάρχουν και άλλοι κανόνες για τις σχέσεις αντρών-γυναικών. Έγινε αναθεώρηση στο Σύνταγμα, ή γίνεται αυτή την εποχή. Έγινε επίσης ε, δημοψήφισμα για να αποφασιστεί η μεταρρύθμιση αυτή του συντάγματος με ιδιαίτερη υψηλή συμμετοχή. Φυσικά και υπάρχουν ακόμα αδυναμίες, αλλά είναι μια χώρα η οποία κάνει τις μεταρρυθμίσεις. Και έτσι λοιπόν θα ήταν κρίμα επειδή οι μεταρρυθμίσεις αυτές γίνονται πιο ήρεμα από τις άλλες χώρες να πούμε ότι δεν γίνονται. Γίνονται. Και το Μαρόκο είναι μια χώρα κλειδί. Και έχει και στην Μεσόγειο ακτές και είναι και κοντά στον Ατλαντικό. Ο Ευχαριστώ. Ο κύριος Παντσέρη από τους σοσιαλιστάς. Δυόμιση λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αντικαθιστώ τον κύριο Γάνκερ που είναι ο αρμόδιος το πρωτόκολλο συμφωνίας με το Μαρόκο δίνει στο Μαρόκο τη δυνατότητα να συμμετέχει στις εργασίες των υπηρεσιών και των άλλων κοινοτικών προγραμμάτων και προβλέπει και τους όρους με τους οποίους μπορεί να συμμετάσχει. Το Μαρόκο δήλωσε ότι ενδιαφέρεται για να συμμετάσχει σε προγράμματα για καινοτομία, ανταγωνισμό και έσαρα Μαρκοπόλο και άλλα. Έτσι δείχνουμε λοιπόν την υποστήριξή μας στις μεταρρυθμίσεις που γίνονται στο Μαρόκο και δίνουμε ένα σημάδι ότι χρειάζεται να συνεχιστούν. Το πρωτόκολλο αυτό ανταποκρίνεται στους νέους στόχους της πολιτικής γειτονίας κείμενο που εγκρίναμε την περασμένη μόλις εβδομάδα στην Αλαμέλεια γιατί είπαμε ότι είμαστε υπέρ της στήριξης των χωρών που εκδημοκρατίζονται αυτή τη στιγμή. Το Μαρόκο έχει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να συμμετάσχει στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και θέλουν και οι δύο πλευρές να ενισχύσουν τη συνεργασία τους γι' αυτό και ο εισηγητής εξ ονόματος της ομάδας των σοσιαλιστών ε, εξέφρασε θετική γνωμοδότηση και είμαστε υπέρ των συμπερασμάτων του. Πρέντα για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να υποστηρίξω την κυρία, να συγχαρώ την κυρία Νέιτ για την εκθεσή της και στη συνέχεια να πω ότι για μας το ΕΛΚ συμφωνούμε απόλυτα με τα συμπεράσματα της έκθεσης, δηλαδή εγκρίνουμε το πρωτόκολλο με το Μαρόκο και όπως η κυρία Νέιτς θα ήθελα και εγώ να τονίσω ότι το πρωτόκολλο αυτό θα επιτρέψει στο Μαρόκο να συμμετάσχει στην εφαρμογή ενωσιακών προγραμμάτων. Θα θεωρείται λοιπόν ισότιμος εταίρος των χωρών μελών θα έχει και κάποια συμμετοχή χρηματοδοτική στα προγράμματα που το ενδιαφέρουν και γι' αυτό νομίζω ότι αυτά που προβλέπει το πρωτόκολλο συμφωνούν και με προηγούμενες συμφωνίες μας με τη χώρα αυτή λόγω δε των αλλαγών που γίνονται εκεί των πολιτικών αλλαγών θα ήταν από εμά η έγκρισή του η ασαφής χειρονομία έγκρισης των μεταρρυθμίσεων. Μετά την απόρριψη από το Κοινοβούλιο του Πρωτοκόλου για την Αλληλεία, θέλουμε τώρα να προτείνουμε τη στήριξη αυτού του πρωτοκόλου γιατί οι Μαροκινοί θα θεωρήσουν τη χειρονομία αυτή ως θετική και ως ενθάρρυνση των μεταρρυθμίσεών τους πολιτικών και οικονομικών. Τέλος, θέλω να αναφέρω ένα λαθάκι που υπάρχει στο τέλος του Σκεπουτικού. Λέει ότι θα γίνουν στις 25 Δεκεμβρίου εκλογές. Όχι, έγιναν στις 25 Νοεμβρίου. 25 Νοεμβρίου, θα γίνουν μάλλον επόμενου Νοεμβρίου ή κυρία Μόνης, Μουνίθ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ευχαριστούμε κύριε Πρέντα, η κυρία Μόνης. Μουνίθ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ απόλυτα με τα όσα είπε η κυρία Νέιτς και τα αναφέρει η σύστασή Θεωρώ ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε το προθυμένο αυτό καθεστώς του Μαρόκου που είναι πολύ σημαντικό, στρατηγική σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να στηρίξει τις επιθυμίες του λαού του Μαρόκου που έχει δεσμευθεί υπέρ πολιτικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων. Αν πραγματικά θέλουμε η ευρωπαϊκή πολιτική γετνίασης να υλοποιηθεί αποτελεσματικά, τότε πρέπει να φροντίσουμε οι διάφορες χώρες να συμμετέχουν στα ευρωπαϊκά προγράμματα υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις βεβαίως που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμμερίζομαι ιδιαίτερα τόσο αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη της κυρίας Νέιτς. Το σημείο στο οποίο αναφέρθηκε και η ίδια για παράδειγμα και που λέει ότι πρέπει ολόκληρη η επικράτεια του Μαρόκο να επωφεληθεί δηλαδή συμπεριλαμβανομένης και της Δυτικής Σαχάρας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για να τηρείται το διεθνές δίκαιο, το οποίο λέει ότι πρέπει από τέτοιε συμφωνίε να υποφελούνται όλες οι περιφέρειες. Εδώ ξέρουμε ότι υπάρχει ένα επίμαχο θέμα. Οι ευρωπαϊκές πολιτικές ε, όμως και εκείνες του Μαρόκου πρέπει να ε, έχουν σαν αποτέλεσμα να υποφελείται από αυτές ολόκληρος ο πληθυσμός της χώρας. Ευχαριστούμε κυρία Γκόμες. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να συγχαρώ την κυρία Νέτς για την έκθεσή της και για τις εξηγήσει της. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι γίνονται μεταρρυθμίσεις στο Μαρόκο. Πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε το το ότι το Μαρόκο είναι στρατηγική σημασίας εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την προηγούμενη εβδομάδα υπερψήφισα την άρση της ελληνικής συμφωνίας με το Μαρόκο, όχι γιατί είμαι κατά μιας ελληνικής συμφωνίας με το Μαρόκο, αλλά γιατί πρέπει οι, οι διαπραγματεύσεις να γίνουν καλά και να λαμβάνουν υπόψη τους το διεθνές δίκαιο όσον αφορά τη Δυτική Σαχάρα. Γι' αυτό και συμφωνώ απόλυτα με τη σύσταση που αναφέρεται εδώ και όπου λέει η κυρία Νέιτς ότι πρέπει να συμμετέχουν όλοι. Δεν πρέπει να το βάζουμε κάτω από το χαλί το θέμα της Δυτικής Σαχάρας. Δεν πρέπει να το κρύβουμε. Αυτοί που το κάνουν δεν είναι πραγματικοί φίλοι του Μαρόκο. Το Μαρόκο έχει ένα πρόβλημα που πρέπει να λύσει και είναι η Δυτική Σαχάρα. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει να κάνει και με την Ευρώπη, γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με το Μαρόκο, πρόκειται για μια περιοχή όπου ακούμε ότι στο Σεχέλ δηλαδή υπάρχουν τρομοκρατικές οργανώσεις. Το ξέρουμε. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να αφήσουμε τη Δυτική Σαχάρα έτσι σε μια κατάσταση η οποία μπορεί να οδηγήσει τους τρομοκράτες να ε, βρεθούν εκεί. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε ένα δυνατό πολιτικό μήνυμα προς τις αρχές του Μαρόκου για αυτό το θέμα. Ευχαριστούμε ο κύριος Βέγγελ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θέλω να συμφωνήσω με τον εισηγητή για την ισορροπημένη του προσέγγιση. Είναι προς το συμφέρον μας η ανάπτυξη καλών σχέσεων με το Μαρόκο. Όπως είπε όμως και ο συνάδελφός μου Γόμες, θέλω επίσης να αναφέρω και το πρόβλημα με την Σαχάρα, τη Δυτική Σαχάρα. Δεν νομίζω ότι ανταποκρίθηκε πολύ σωστά το Μαρόκο με τον αλλιευτικό πόλεμο κατά της Ένωσης αμέσως μετά αυτά που έγιναν την περασμένη εβδομάδα στο Κοινοβούλιο. Φυσικά υπάρχουν σοβαροί λόγοι, αλλά πρέπει να καταλάβει το Μαρόκο τι εννοούσε η χειρονομία μας αυτή εφόσον μάλιστα έχει νεοεκλεγέν καινοβούλιο. Επισκέφθηκα πρόσφατα τη Δυτική Ζαχάρα και κατάλαβα ότι ο πληθυσμός της που ζει σε αντίσκηνα και στρατόπεδα δεν ωφελείται από καμία συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή με, από τη συνεργασία Ένωσης και Μαρόκου πρέπει να βρεθεί μια λύση στα Ηνωμένα Έθνη με δημοψήφισμα. Η προετοιμασία του δημοψηφίσματος έγινε. Όπου το Πολυσάριο συνεργάστηκε με την κυβέρνηση του Μαρόκου. Το θέμα λοιπόν είναι απλώς να ληφθεί η πολιτική απόφαση. Καλά θα έκανε νομίζω το Μαρόκο να εφαρμόσει αυτά που ζήτησε η διεθνής Κενότης. Δηλαδή να οργανωθεί το δημοψήφισμα και να πάψει ο διωγμός του λαού της Δυτικής Σαχάρας. Ευχαριστούμε ο κύριος Αρλάκη. Ευχαριστώ και εγώ συμφωνώ με τους συναδέλφους. είναι θετικό, θετική η συμφωνία αυτή. Θέλω να πω δύο σχόλια. Πρώτον, πρέπει να υποστηρίξουμε τις δυνάμεις που αγωνίζονται στο Μαρόκο για τη δημοκρατία. Ταυτόχρονα όμως δεν πρέπει να θεωρούμε, τη θεωρούμε τη διαδικασία αυτή ως δεδομένη. Μέχρι τώρα είδαμε ότι υπάρχει μία μεταρρυθμιστική πρόθεση ή τάση, αλλά στην πράξη πολύ λίγα είδαμε. Οι μεταρρυθμίσεις που έγιναν μέχρι τώρα ήταν αρκετά αδύναμες. Δεν έχει γίνει ούτε δημοκρατία, ούτε κοινοβουλευτική μοναρχία το Μαρόκο. Το πρόβλημα της Δυτικής Σαχάρας το λέει αρκετά το έγγραφο. Θα θέλαμε το Μαρόκο οι συμφωνίες μας με το Μαρόκο να ωφελούν και το λαό της Δυτικής Σαχάρας. Πρέπει όμως να τονίσουμε πολύ σαφέστερα από ό,τι πριν ότι η Δυτική Σαχάρα δεν είναι τμήμα του Μαρόκου. Και οποιαδήποτε συμφωνία δεν το αναγνωρίζει αυτό δεν είναι σωστή συμφωνία και παραβιάζει τις ίδιες τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμφωνώ λοιπόν βασικά με όλα, αλλά θα ήμουν ακόμη πιο ικανοποιημένος αν αυτές οι αρχές εκφράζονταν σαφέστερα. Τώρα η κυρία Νέιτς για τα συμπεράσματά της. Κυρία Πρόεδρε, να με συγχωρήσουν οι συνάδελφοι, αλλά δεν θέλω τώρα να μπω στις λεπτομέρειες για τη Δυτική Σαχάρα, γιατί θεώρησα απαραίτητο μεν να το αναφέρω, γιατί είναι θέμα τριβών με την κυβέρνηση του Μαρόκου, πρέπει να συνεχίσουμε να το προσέχουμε. Έχω και εγώ μια άποψη, αλλά δεν έχει καμία σχέση με το θέμα μας εδώ. Ευχαριστώ τους συναδέλφους που μίλησαν εξ ονόματος των ομάδων για το ενδιαφέρον τους για το θέμα μου και για την έγκριση του πρατακόλου που είναι όντως πολύ σημαντικό. Επί ενός θέματος θέλω να επανόλθω αυτού που είπε ο κύριος Αρλάκης για την πρόταση που συμπεριλαμβάνεται στην ε, συνταγματική μεταρρύθμιση στο Μαρόκο. Είναι πολύ λεπτό θέμα για υπηκόους ε, συνταγματικής μοναρχίας να επικρίνουν άλλες συνταγματικές μοναρχίες. Εγώ νομίζω ότι οι μεταρρυθμίσεις που προτείνονται στο Μαρόκο είναι πολύ σημαντικές. Πρέπει βέβαια να δοκιμαστούν στην πράξη, αλλά ίσως οι συνάδελφοι που δεν γνωρίζουν καλά την κατάσταση στο Μαρόκο ξέχασαν κάτι. Απαγορεύεται στο Μαρόκο να αλλάξει η πολιτική σύνθεση μιας βουλής κατά τη θητεία της. Υπάρχουν κόμματα που απαγορεύεται η ίδρυση κομμάτων κατά τη διάρκεια μιας θητείας. Αυτό που επιτρέπεται είναι ότι ξαφνικά ξεφυτρώνουν διάφορα κόμματα αμέσως πριν τις εκλογές και μετά εξαφανίζονται μετά. Τέλο πάντων, το σημαντικό είναι ότι υπάρχει πλουραλισμός, πολλαπλά πολιτικά κόμματα με ιστορία που παίρνουν μέρος σε εσωτερική συζήτηση σε με σημαντικό βαθμό. Υπάρχει αυτή τη στιγμή δημιουργείται μία κυβέρνηση συνασυπισμού και είναι τα πράγματα λίγο καλύτερα από ό,τι γειτονικέ χώρες μέχρι στιγμής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Υπενθυμίζω ότι η διορία κατάθεση τροπολογιών λήγει στις 10 Ιανουαρίου το μεσημέρι. Συνάδελφοι, τώρα το σημείο 7 της ημερήσιας διάταξης, η ανταλλαγή απόψεων για το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την έκθεση περί της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Ο κύριος Βίτο εισηγητής έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και καλημέρα σε όλους. Ε, γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που έχω την τιμή και τη χαρά να παρουσιάσω μια έκθεση για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Ε, φέτος ορίστηκα εισηγητής και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους στην Επιτροπή Συμπεριλαμβανομένων και των Σκιωδών με τους οποίους συναντήθηκα και προσπάθησα να ε, σφυριλατήσω ευθύ εξ αρχής σε μια καλή σχέση. Ε, να συμπεριλάβω τις απόψεις τους ε, έτσι ώστε η έκθεσή μου να εγκριθεί από το Κοινοβούλιο. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και όλους εκείνους που βρίσκονται στη χώρα την ίδια είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ τη χώρα, όχι μόνο τα Σκόπια, αλλά ολόκληρα τη χώρα, σε πέντε διαφορετικές ε, περιπτώσεις. Πήγα και ιδιωτικά ε, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου των εκλογών και είδα πόσο επιτυχής ήταν η διεξαγωγή των εκλογών. Μπόρεσα να μιλήσω ε, στην δεκαετή επέτειο για την ενδιάμεση συμφωνία προσεκλήθη να μιλήσω σε μια συνάντηση που έλαβε χώρα στα Σκόπια και μίλησαν Υπουργείο Εξωτερικών όλων των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Συναντήθηκα και με νέους ε, από όλα τα Δυτικά Βαλκάνια, όχι μόνο από τη χώρα αυτή, ε, με θέμα την αντιμετώπιση του ρατσισμού και την δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης. Αυτό έλαβε χώρα στην λίμνη της ε, Οχρίδας, ε, πολύ συμβολικό το μέρος και ελπίζω ότι μπόρεσα να συμμετέχω επικοδομητικά στην τελευταία συνάντηση της ε, Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις ήμουν ιδιαίτερα ευπρόσδεκτος, παρότι βέβαια όσον αφορά την διαδικασία της Διεύνησης Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν και πάρα πολλά πολιτικά στοιχεία που εμπλέκονται. Συζητήθηκαν αυτά σήμερα το πρωί. Πολλές φορές ξεχνάμε ότι μιλάμε εδώ για μια χώρα, ε, για ένα λαό, ιστορία, πολιτισμό. Θέλω λοιπόν να πω ότι χάρηκα ιδιαίτερα που ε, γνώρισα αυτή τη χώρα, την κοινωνία της και ε, αισθάνομαι ακόμα πιο ενθουσιασμένος όσον αφορά στις προσπάθειές μου για την ένταξη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ καλύτερα τώρα από ότι όταν ήμουνα από όταν πρωτοδιορίστηκα στην αρχή εισηγητής. Λοιπόν, ως εισηγητής εγώ προσπάθησα να βασιστώ σε παλαιότερες εκθέσεις. Ε, σε κάποια στοιχεία της έκθεσής μου υπάρχουν ε, χωρία τα οποία έχω υιοθετήσει από παλαιότερες εκθέσεις. Όσοι με γνωρίζουν, γνωρίζουν πολύ καλά ότι έχω και εγώ τη δική μου την προσωπική προσέγγιση, έχω τη δική μου προσωπικότητα και επειδή μου δόθηκε η τιμή να είμαι εισηγητής για αυτό το θέμα, θέλησα και εγώ να αφήσω το δικό μου το αποτύπωμα. Έτσι λοιπόν σε αυτό το σχέδιο έκθεσης προσπάθησα σε αρκετά σημεία να προβάλλω αυτό που σας είπα, να δώσω την προσωπική μου νότα. Καταρχήν, όσον αφορά στο σχέδιο, ε, η παράγραφος 1, ε, η πρόταση υπαριθμών 1, εκεί υπάρχει μια σαφέστατη δήλωση ότι θέλουμε να υπάρχει μια συγκεκριμένη ημερομηνία για τις ε, συζητήσεις χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση. Αυτή είναι η θέση του Κοινοβουλίου, αλλά θέλω να το καταστήσω ε, περισσότερο σαφές εκπέμποντας μήνυμα τόσο στις Βρυξέλλες όσο και στη χώρα την ίδια και σε ολόκληρη την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό αφορά παράγραφο 1, πρώτη πρόταση. Επίσης, θέλησα να εξετάσω μία σειρά εναλλακτικών λύσεων για να προχωρήσουμε χωρί ε, προκαταλήψει αναζήτησα μια εναλλακτική λύση και κοίταξα τις δυνατότητες που υπάρχουν. Κυρίως ε, ε, είδα τις εκθέσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής είδα ε, τι, προτείνει, ε, τι προέτεινε εδώ ο Υπουργό Εξωτερικών κ. Ποπόφσκι πριν από ένα μήνα που είπε ότι θα πρέπει να οριστεί μια συγκεκριμένη ημερομηνία έτσι ώστε να ε, διευθετηθεί και το διμερές πρόβλημα. Εγώ ε, και πάλι προβάλλω αυτή την εναλλακτική λύση με στόχο να περάσουμε στη δεύτερη φάση της σταθεροποίησης και της διαδικασίας ε, προσχώρησης. Ε, σας λέω ότι αυτό χωρίς καμία προκατάληψη για τις συζητήσεις που κατά άποψή μου πρέπει να ξεκινήσουν. Γι' αυτό εξέτασα τι εναλλακτικέ λύσει. Να πω επίση ότι το status quo, η διατήρηση των κεκτημένων, δεν είναι εναλλακτική λύση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, πάντα αυτά που λέει ακούγονται και στην χώρα αυτή ιδιαίτερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι θετική ε, βέβαια αυτό δεν είναι θέσφατο όπως αναφέρεται στην έκθεση εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας δεν μπορούμε να τη θεωρούμε ούτε και αυτή δεδομένη. Έχω ένα μεγάλο κομμάτι ε, για την οικονομική ανάπτυξη και εκεί φαίνεται πως ε, τα ε, πηγαίνει μια χαρά η χώρα σε θέματα μακροοικονομικής ανάπτυξης, σταθερότητας. Γι' αυτό πρέπει να τους επενέσουμε και γι' αυτό το αναφέρω στην έκθεση. Βεβαίως ασκώ και έντονη κριτική για θέματα μεταρρυθμίσεων. Όμως ε, το κάνω αυτό, ελπίζω, ε, κάνοντας σχόλια που είναι σαφή έτσι ώστε όσοι θέλουν μεταρρυθμίσεις ε, στη χώρα να δούνε τι προβλήματα υπάρχουν. Και τα κάνω αυτά με επικοδομητικό ύφο γλώσσας, γιατί θέλω να αποδείξω στου πολίτες της χώρας ότι οι συστάσεις, οι προτροπές οι δικές μας ε, δεν σημαίνουν ότι θέλουμε να ξεφύγουμε από την αμοιβαία επιτιμία να στεφτεί το εγχείρημα από επιτυχία. Εγώ απευθύνομαι όχι σε πολιτικούς, αλλά και σε άλλα στελέχη της πολιτικής, ε, απευθύνομαι στην κοινωνία των πολιτών. Δεν θέλησα να να συναντήσω μόνο πολιτικού, αλλά να συναντήσω και απλού πολίτες. Γι' αυτό λοιπόν καλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενισχύσει σε μεγάλο βαθμό αυτό το εργαλείο της κοινωνίας των πολιτών. Μερικοί είπαν ότι δεν θα έπρεπε να το κάνω αυτό, γιατί αυτό είναι σχέδιο κοινοβουλευτικού ψηφίσματος. Γιατί να μην τους ε, συγχαρώ που τα πήγανε καλά στο μπάσκετ, ε, στο πρωτάθλημα του μπάσκετ. Αυτά είναι σημαντικά για τους ανθρώπους επιτόπου. Είδα πως γιόρτασαν και πιστεύω ότι πρέπει να συμμεριζόμαστε τα συναισθήματα των πολιτών, έτσι θα τους φέρουμε πιο κοντά μας. Και λέω με απόλυτα σαφήνεια ότι η απελευθέρωση των θεωρήσεων είναι ε, καθοριστικό στοιχείο των σχέσεών μα. Και εδώ στο Κοινοβούλιο θα το υπερασπιστούμε. Τώρα, στο θέμα της ε, ονομασίας, να πω το εξή. Εγώ δεν προσπαθώ να είμαι ο διαμεσολαβητής, έχουμε διαμεσολαβητή στα Ηνωμένα Έθνη. Εγώ προσπάθησα να ε, κατεβάσω τις ε, προσδοκίες και όσον αφορά το ρόλο μου του εισηγητή. Δεν είναι δική μου δουλειά να λύσω το θέμα της ονομασίας και πιστεύω αν προσπαθούσα να το κάνω αυτό, τότε θα προκαλούσα περισσότερη ζημιά από καλό. Αυτό που προσπάθησα και προσπαθώ να κάνω σε αυτήν την έκθεση είναι να ασκήσω πίεση, επικοδομητική πίεση σε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές και στην Αθήνα και στα Σκόπια για να υπάρξει μια δίκαιη συμφωνία που θα είναι δίκαιη αποδεκτή και για τις δύο πλευρές. Νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη θέση που εγώ μπορώ να λάβω. Και γι' αυτό έχω υιοθετήσει πολλά χωρία από ε, παλαιότερες ε, εκθέσεις που μπλοκάρισαν την πρόοδο της χώρας και της ε, διαδικασίας ένταξης. Είναι σημαντικό να υπάρχουν καλές γειτονικές σχέσεις. Καλό την Επιτροπή να καταθέσει ε, έναν μηχανισμό διαιτησίας ευρέως αποδεκτό για διμερείς ε, αντιπαραθέσεις, όχι μόνο εδώ, αλλά γενικότερα για όλη τη διαδικασία διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαφορά τώρα σε σχέση με την περίπτωση αυτή είναι η εξής. Εγώ αναφέρω την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, του Διεθνούς Δικαστηρίου. Θα ήταν σημαντικό να ληφθεί μια απόφαση χωρίς αυτήν την απόφαση. Υπάρχει όμως τώρα η απόφαση και ζήτησα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πούν ποια είναι η δική τους η σύσταση μετά την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης. Δεύτερον, εγώ δεν θα πω στην Ευρωπαϊκή Ένωση να λύσει το θέμα, αλλά όταν θα λυθεί το θέμα δίκαια, δεν πρέπει να το στοπουλήσουμε. Θα υπάρξει δημοψήφισμα. Εμείς πρέπει να ρίξουμε το βάρος μας σε αυτή την ε, εκστρατεία του δημοψηφίσματος. Να πω επίσης τρίτον ότι αν η χώρα καταφέρει να επιτύχει και άλλες μεταρρυθμίσεις, εγώ πιστεύω ότι αυτό από μόνο του θα βοηθήσει έτσι ώστε το περιβάλλον, η περιραίουσα ατμόσφαιρα να διευκολύνει την επίλυση του προβλήματος. Τέταρτον, χρησιμοποιώ τη λέξη Μακεδονία. Τη χρησιμοποιώ μία φορά αλλά τη χρησιμοποιώ με απόλυτη σαφήνεια στην παράγραφα υπαριθμών 8. Αυτή ήταν η θέση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν χρησιμοποιώ με τη λέξη Μακεδονία, αλλά μακεδονικό, ω επίθετο. Αυτό το έκανε η Επιτροπή και φέτος πολλοί διαπίστωσαν ότι στη χώρα αυτή έγινε μεγάλο θέμα το να μην χρησιμοποιείται το επίθετο μακεδονικός σε σχέση με τον πολιτισμό τους, τη γλώσσα τους και την ταυτότητά τους, αυτό είχε ιδιαίτερα αρνητική απήχηση κυρίως όταν ε, δημοσιεύτηκε η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή είναι και η πρακτική που ισχύει στα Ηνωμένα Έθνη. Είναι απόλυτα συνεπής και με την ε, απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Το επίθετο αυτό το μακεδονικό δεν το βάζω για να προκαλέσω κανένα, αλλά πρέπει να δείξουμε ότι εισπράξαμε το μήνυμα της χώρας, την αντίδρασή της. Άκουσα πολύ προσεκτικά την Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή όταν διαπραγματεύτηκαν το κείμενο στην συνάντηση και τους είπα ότι αν τελικά μπορέσουν να καταλήξουν σε μια συμφωνία ε, και το έκαναν, τότε και εγώ θα έπρεπε να το κάνω το ίδιο στην δική μου την έκθεση. Έτσι λοιπόν με τη σύνταξη αυτής της έκθεσης αυτό θέλησα να κάνω. Αυτά που σας παρουσιάζω είναι και λιγότερα από αυτά που συμφωνήθηκαν στην Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή. αυτοί χρησιμοποιούν τη λέξη «expact». Εγώ χρησιμοποιώ πιο ευγενικό ύφο. Νομίζω δεν έχουμε πλέον χρόνο στη διάθεσή μας. Δεν θα αναφερθώ σε άλλες προτάσεις για μεταρρυθμίσεις. Θα ακούσω πολύ προσεκτικά αυτά που έχουν να πούν οι υπόλοιποι συνάδελφοι και θα κάνω ό,τι μπορώ για να απαντήσω. Να πω όμως το εξή σε εσά, στους συναδέλφους μας. Το status quo δεν είναι εναλλακτική λύση. Χαίρομαι για την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο Μαυροβούνι, στη Σερβία. Ε, χαίρομαι ιδιαίτερα που θα ενταχθεί η Κροατία. Εγώ όμως είμαι ο εισηγητής σας για την πρώην δημοκρατική δημοκρατία της Ιουγκοσλαβίας στη Μακεδονία και πρέπει να πω ότι δεν πρέπει να το ξεχάσουμε το θέμα. Και αν το ξεχάσουμε, εγώ σας επισημαίνω ότι θα υπάρχουν επιπτώσεις στις διεθνωτικές σχέσεις στη χώρα, επιπτώσεις στην περιφερειακή σταθερότητα και επιπτώσεις στην ίδια τη διαδικασία διεύρυνσης. Έτσι λοιπόν το Συμβούλιο τον Μάρτιο όταν θα επανεξετάσει το θέμα της διεύρυνσης επιθυμώ να λάβει υπόψη του και την χώρα αυτή. Και στο ψήφισμά μας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αυτό θα ζητήσω από το Συμβούλιο να πράξει. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Χουίτ. Έξι ζήτησαν το λόγο αλλά μετά θα ψηφίσουμε. Γι' αυτό παρακαλώ να είστε πολύ σύντομοι, Εφτά μάλλον, ο κύριος Κόβατς εκ πρώτος και καλύτερος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Χόουιτ για την πρόταση του. Την πρόταση αυτή αναφέρονται όλα τα σημαντικά στοιχεία. Εμείς ε, θέλουμε το θέμα αυτό να το διαχωρίσουμε κάπως από την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, αλλά δεν είναι δυνατόν, γιατί μόνο στο πλαίσιο της προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δυνατόν να επιληθούν και τα προβλήματα του παρελθόντος. Στο ιστά ψηφίσματά μας ε, έχουμε προτείνει να υπάρξουν, να οικοδομηθούν ε, γέφυρες εμπιστοσύνη με τις γειτονικές χώρες και νομίζω ότι αυτό είναι μια πολύ καλή πρόταση και σε σχέση με τη Μακεδονία. Δυστυχώς τα γεγονότα είναι διαφορετικά εν της πράγμαση. Δεν υπάρχει πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά ε, κάποιες ε, ημέρες εορτασμού της ε, Μακεδονίας και της Βουλγαρίας. Στη Μακεδονία έχουμε βιβλία που υποδαβλίζουν το μίσος κατά της Βουλγαρίας η Μακεδονία είναι η μόνη χώρα που προχωράει με αρνητική ταυτότητα. Οι Μακεδόνες λένε είμαστε Μακεδόνες γιατί δεν είμαστε Βούλγαροι. Το αίσθημα της εθνικής ταυτότητας ε, και του πολιτισμού είναι θέμα ε, κράτους, του κράτους, αλλά όμως αυτό εμείς δεν μπορούμε να το ανεχτούμε. Δεν μπορούμε να παραμένουμε αντρανείς και να μην κάνουμε τίποτα. Δεν έχουμε καμία αντίρρηση οι Μακεδόνες να αποκαλούνται Μακεδόνες. Έχουμε όμως κοινή ιστορία και αυτή πρέπει να γίνεται σεβαστή. Το ίδιο ισχύει και για τις ε, εκφράσεις και λέξεις μίσους που απορρέουν από την πρώην γιουγκοσλαβική γλώσσα. Ελπίζω λοιπόν οι εταίροι μας στην ε, Μακεδονία να αποστασιοποιηθούν από το παρελθόν τους και να στραφούν προς ένα κοινό ευρωπαϊκό μέλλον. Ευχαριστούμε. Όχι πάνω από 1,5 λεπτό. Παρακαλώ, κύριε Βεργκίν. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομος. Πρώτα απ' όλα, συγχαρητήρια στον κύριο Χόουιτ για το έργο του. Ιδιαίτερα μάλιστα μετά τα τελευταία γεγονότα έπρεπε πολύ γρήγορα να προχωρήσει σε αυτό το θέμα. Έκανε όμως πολλές προσπάθειες για να μάθει περισσότερα πράγματα για την Μακεδονία, να ενημερωθεί και να φροντίσει για την έκθεση αυτή που αναφέρεται στις σχέσεις μας. Όπω είπε και αυτό πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να βγούμε από τα διέξοδο. Η κατάσταση μέσα στη χώρα επιδεινώνεται για διαφορετικούς λόγους, αλλά ένα από αυτού είναι ότι η χώρα δεν μπορεί να ξεκινήσει τι διαπραγματεύσει ή τέλο πάντων βρίσκεται σε αδιέξοδο όσον αφορά την πορεία τη προ την Ευρωπαϊκή Ένωση για τρίτη στη συνέχεια χώρα. Για τρίτη φορά, για τρίτη φορά επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι δεν μπορούν να προχωρήσουν οι συνομιλίες. Φυσικά και υπάρχουν ευαισθησίε για αυτό το θέμα από την ελληνική πλευρά, αλλά πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη μας και τη δύσκολη κατάσταση μέσα στην οποία βρίσκεται και η Μακεδονία. Φυσικά δεν είμαστε ένα κοινοβούλιο που μπορεί να διαπραγματευτεί ή τέλο πάντων να μπορεί να βρει λύσεις. Όλα βρίσκονται στα χέρια των κυβερνήσεων των δύο πλευρών. Χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι δεν μπορούμε κι εμείς να δώσουμε κάποιες ιδέες για τις εξελίξεις όσον αφορά τις σχέσεις αυτές. Θεωρούμε ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή κυβερνητικά σώματα λαμβάνοντας υπόψη τις πρωτοβουλίες της ε, ε κυβέρνηση της Μακεδονίας, αλλά λαμβάνοντας υπόψη επίσης και την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα, να αρχίσουν και πάλι οι συνομιλίες για αυτό το θέμα. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, τα πολιτικά μηνύματα που έρχονται από τη Μακεδονία συχνά είναι αρνητικά απέναντι σε γείτονες χώρες τους, αλλά πρέπει να μεταφέρουμε το μήνυμα εδώ ότι δεν περικυκλώνεται από εχθρούς η Μακεδονία, ότι νοιαζόμαστε για τη χώρα αυτή. Αυτή η ψυχολογική προσέγγιση πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει. Ευχαριστούμε κύριο Κασουλίδης. Merci, Madame. Ευχαριστώ. κυρία μου. Συγχαίρω και εγώ τον κύριο Χάουιτ και θέλω να προσθέσω ότι έβαλε στο σωστό πλαίσιο τον ρόλο του Κοινοβουλίου. Δηλαδή είπε ότι όλοι θέλουν η ΦΥΡΟΜ να αρχίσει διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση για ένταξη χωρίς καθυστερήσεις. εφόσον υπάρχουν οι συνθήκες. Και δέχομαι το πνεύμα με το οποίο παρουσίασε, με το οποίο εννοεί το ρόλο του Κοινοβουλίου στη διαμάχη της ονομασίας, όπως φαίνεται στην παράγραφο 7. θα ήθελα να του ζητήσω να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο διατυπώνει την παράγραφο 9. Γιατί η θέση μας είναι ότι όσο πιο πολλές προϋποθέσεις τίθενται από τις δύο πλευρές, τόσο, όσο πιο πολλοί όροι, τόσο δυσκολότερο γίνεται να λυθεί η διαμάχη και σε αυτή την περίπτωση θέλουμε να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις όσο το δυνατόν νωρίτερο να τεθεί διορία για την επίλυση της ε, διαφοράς της ονομασίας είναι κάτι που δεν θα διευκολύνει τη λύση. Ως προς την ιδέα του δε συνταγματικής αλλαγής ώστε ο μηχανισμός διαμεσολάβησης, να, ώστε να χρησιμοποιηθεί ένας μηχανισμός με διαμεσολάβηση, δεν ξέρω αν είναι ρεαλιστικό κάτι τέτοιο. Τότε γιατί να μην έχουμε διαπραγμάτευση και στις διαφορές μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και υπολείπων χωρών της Ένωσης. Κυρία Κοπά. Uh, και εγώ θέλω να συγχαρώ τον κύριο Χόβιτ για το τόσο ισορροπημένο κείμενό του και για τις προσπάθειες που έκανε να καταλήξει σε ένα κείμενο μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Βρίσκω πολύ ενδιαφέρουσα και τη νέα μορφή, την παρουσίαση του συγητή. Πιστεύω ότι δίνει περισσότερο, μεγαλύτερο δυναμισμό και δείχνει πιο ξεκάθαρα τα θέματα τα οποία έχει να αντιμετωπίσει η χώρα. Τρία σύντομα σημεία. Αυτό που λείπει για μένα στο κείμενο είναι κάποια μνήα που σε παλιότερες εκθέσεις είχαμε βάλει για antiquization. Δημιουργούνται πολλά αρνητικά συναισθήματα απέναντι στη χώρα και είναι κάτι που συνδυάζεται και με αυτό που ανέφερε ο συνάδελφος Κόβατσεφς με το μίσος. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό το χαρακτηριστικό της κυβέρνησης δεν βοηθάει τις διαπραγματεύσεις ούτε την αμοιβαία κατανόηση. Δεύτερον, Δεύτερον. το status quo δεν αποτελεί επιλογή για την περιοχή. Ναι, συμφωνώ. Αλλά αυτό αποφάσισε το Συμβούλιο. να σκεφτούμε και την ε, Σερβία και το Μαυροβούνι. Και αυτό το οποίο αποφάσισε πριν από μερικές μέρες το Συμβούλιο είναι να διατηρήσει το στάτος κουβό. Τελευταίο σημείο. Έχετε απόλυτο δίκιο ότι πολλές φορές ο εισηγητής και όχι μόνο για την περίπτωση της Φύρωμα αλλά και για άλλες προς χώρες προσπάθησε να παίξει τον ρόλο του διαμεσολαβητή και αυτό είναι λάθος. Δεν βοηθάει και ε, οδηγεί στα αντίθετα αποτελέσματα. Αυτά ευχαριστώ πολύ και θα έχουμε την ευκαιρία της καλλιώς να επανέλθουμε και αργότερα πάνω στο κείμενο. Ο κύριος Νικολάη. Ευχαριστώ. Δύο πράγματα θέλω να πω εγώ. Η ελευθερία τύπου. τύπου. Είναι κάτι που πρέπει να αναφερθεί στην έκθεση. Γιατί έχουμε κάποια προβλήματα αυτή τη στιγμή στην ε, Μακεδονία. Και για τη Μακεδονία και για μας είναι η απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη στα πλαίσια ε, της ε, ενέργειας της Ελλάδας να μπλοκάρει την ε, χώρα. Πρέπει να συμμορφωθούμε προς μια νομική απόφαση ή όχι. Έπειτα υπάρχει το θέμα των μειονοτήτων. Υπάρχει πρόοδος στην Μακεδονία για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται το θέμα, αλλά σίγουρα πολλά μπορούν να γίνουν ακόμα για να τηρούνται πλήρως τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Κορνέλισεν. Θέλω κι εγώ ε. να συγχαρώ τον κύριο Χόβιτ για την τόσο καλή του έκθεση. Και μου αρέσει το σημείο 10 που αναφέρεται στην ε, έκθεση. Είναι κάτι που το θέλαμε και εμείς. Και εμείς. Δεν είναι θέμα βέβαια μόνο διμερές. Νομίζω ότι εμείς ως νιόριμη πολιτική ένωση πρέπει να έχουμε τρόπο να το λύσουμε και να βρούμε μια λύση αντί να αφήνουμε τη χώρα αυτή να είναι μπλοκαρισμένη όσον αφορά την πρόσβασή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είδα επίσης ότι δίνεται πολύ προσοχή στο θέμα του ε, σεξουαλικού προσανατολισμού, την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Για το πρώτο θέμα βλέπω ότι γίνονται διάφορα στην ε, νομοθεσία. Πρέπει πράγματι να αλλάξει η νομοθεσία της χώρας για τα θέματα αυτά. Και ελπίζω ότι θα το κάνει αυτό γρήγορα. Τέλος, για την μειονότητα στην Αλβανία. Τα τελευταία θέματα που έχουν προκύψει στο Κωσυφοπαίδιο έχουν περάσει και στη Μακεδονία. Και αντί να υπάρχει ηρεμία, δυστυχώς διαπιστώνουμε ε, περισσότερη σύγχυση και προβλήματα. Ίσως θα ήταν καλό να αναφέρεται αυτό στην έκθεση. Τώρα κάποιες τροπολογίες θα υποβάλουμε και εμείς, αλλά γενικά μιλώντας, όπως σας είπα, είμαστε ευχαριστημένοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριο Στάνοκ. Uh, Ευχαριστώ. Εγώ συγχαίρω τον κύριο Χάουιτ. Ιδιαίτερα μου ήρεσε η παράγραφος όπου συγχαίρει τη Μακεδονία γιατί κέρδισε στο μπάσκετ ενώ έπαιζε και η Ελλάδα. Λυπούμαστε όμως για την απόφαση του Συμβουλίου να μπλοκαριστεί η συνέχεια των ενταξιακών διαπραγματεύσεων γιατί η πρόσφατη απόφαση από το Διεθνές Δικαστήριο για το θέμα της υποψηφιότητάς της στο ΝΑΤΟ λέει πολλά και για τις υποχρεώσεις που έχει διεθνώς η Ελλάδα. Ελπίζω όλα αυτά να ενθαρρύνουν την Αθήνα να λύσει το πρόβλημα της ονομασίας και να μην εμποδίζει τη Μακεδονία από το δικαίωμά της να μπει στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Δεν υπάρχει καμία δικαιολόγηση για την συνέχιση της παρεμπόδισης αυτής είναι, ευημερούν και ανεξάρτητο κράτος και κοινωνία που έχει αρκετά λεπτά προβλήματα. Πρέπει λοιπόν να υποστηρίξουμε την πολυπολιτισμική, τον πολυπολιτισμικό της χαρακτήρα και να μην την κρατάμε απομονωμένη 6-7 χρόνια χωρίς δικαίωμα να προχωρήσει στην επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων και αργά ή γρήγορα θα τους αποστεθεροποιήσει αυτό. Πρέπει απειγόντως να βρούμε τρόπους να βελτιωθεί αυτό μέχρι την επόμενη σύνοδο. Οι συντηρητικοί είναι πολύ φίλοι της Μακεδονίας και θα παραμείνουν τέτοιοι. Ευχαριστώ κυρία μου συγχαίρω και εγώ τον κύριο Χόουιτ επειδή δεν έχουμε χρόνο θα επιμείνω μόνο στην παράγραφο 22. Και εμείς είμαστε υπέρ της έναρξης των διαπραγματεύσεων γιατί αυτό συμφέρει όλους. Αλλά θέλω να προσθέσω ότι οι ιστορικές διαφορές που συνδέονται με αυτή τη διαδικασία πρέπει να προσέξουμε και την ερμηνεία των ιστορικών γεγονότων. Στην παράγραφο 22 πρέπει να δούμε αυτό το θέμα των σχολικών βιβλίων. Έχω δει φοβερά παραδείγματα έκφρασης μίσους προς γειτονικέ χώρες. Και αυτό όχι μόνο σε εθνοτική βάση, αλλά είναι πολιτικό. Υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα. Μικτές επιτροπές λοιπόν ή και συνέδρια για τα ιστορικά θέματα είναι κάτι που είναι τελείως απαραίτητο. Θα ήθελα να πω ότι φυσικά μερικοί θύνοντες του μακεδονικού κράτους λένε αυτά θα τα διορθώσουμε όταν θα μπούμε. Μπορεί όντως κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων να δημιουργηθούν οι καλύτερες συνθήκες για καλή γειτονία. Ο κύριος Πέτερλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ δεν χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί συνεχίζεται αυτή η πολύπλοκη διαμάχη μεταξύ των δύο χωρών της Ελλάδας και της Μακεδονίας. Βλέπω ότι χρησιμοποιούνται πολλά και διαφορετικά ονόματα για την ίδια χώρα και αυτό την εμποδίζει να προχωρήσει. Μερικές φορές δεν αναφέρεται καν το όνομα της χώρας. Άλλες φορές οι συζητήσεις μοιάζουν με το πρόβλημα της κότας και του αυγού. Συμφωνώ ότι αυτό που πρέπει να γίνει τώρα είναι να βρεθεί ένας επικοδομητικός τρόπος για να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει πρώτα να υπάρχει αμοιβαίως σεβασμός και των ταυτοτήτων του καθενός. γιατί εδώ αμφισβητείται η ίδια η ταυτότητα της μιας χώρας, ακόμη και της γλώσσας της. Αυτό το είπα όταν άκουσα ότι υπάρχει αυτή η τάση να μην χρησιμοποιείται το επίθετο μακεντόνσκι για τη γλώσσα. Νομίζω ότι από τότε τα πράγματα χειροτέρεψαν κιόλας. Δεν ξέρω πώς θα αισθανόμουν ο ίδιος αν κάποιος μου έλεγε ότι δεν μπορώ να ονομάζομαι πια Σλοβαίνος ή ότι πρέπει να ψάξω στην ιστορία άλλο όνομα που είχε ο λαός μου. Πολλές φορές υπόθηκε εδώ ότι πρέπει να σεβόμαστε την ιστορία αλλά δεν νομίζω ότι είναι σωστό να πηγαίνουμε τόσο παλιά πίσω για να ψάχνουμε με το ζόρι λύσεις. Εγώ θα ήθελα οι γείτονε να συνομιλούν και να συμφωνούν για αυτά τα θέματα και να υπάρχει πρόοδος με αμοιβαίο σεβασμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ολοκληρώνουμε αυτό το θέμα. Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών είναι η 10η Ιανουαρίου στις 12 το μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βόβιτς. Τώρα θα περάσουμε στις ψηφοφορίες παρακαλώ. Κύριε Σάριος Βολσκιά δεν είναι εδώ ακόμα. Οπότε θα ξεκινήσουμε με την έκθεση του κυρίου Βάτσον. Θα ψηφίσουμε πρώτα την κυρία Βάτσον. Πρόκειται για το σχέδιο έκθεση περί πρώτα σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προ το Συμβούλιο σχετικά με μια συνεκτική πολιτική έναντι των αυταρχικών καθεστώτων κατά των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει περιοριστικά μέτρα όταν αυτά προωθούν τα προσωπικά και εμπορικά του συμφέροντα εντό των συνόρων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχετε τι ε, ηλεκτρονικέ σα κάρτε για την ψηφοφορία. Ωραία, ξεκινάμε. Τροπολογία 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα επαληθεύσουμε. Διότι δεν είναι ξεκάθαρο το αποτέλεσμα. Τροπολογία 36 λοιπόν. Ε, Επαληθεύουμε ναι. ηλεκτρονικά παρακαλώ. Τελειώσατε. Ψηφίσατε. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 4. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 39, υπέρ, κατά, αποχές, οι σοσιαλιστές δεν ψηφίζουν, καλό θα ήταν να συμμετέχουν και εκείνοι στην ψηφοφορία μια που είναι εδώ, εγκρίνεται. Μια στιγμή, μια στιγμή, δεν ξέρω τι θα κάνουν. Ξανά, τροπολογία 39, υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 50 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 52 υπέρ, κατά, αποχές θα επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία 52. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα της ψηφοφορίας. Κύριε Σάριους Βόλσκι. απορρίπτεται. Απορρίπτεται. 53 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 54 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 59. Έχει αποσυρθεί όμως. Οπότε περνάμε στην τροπολογία 63. Δίνω το λόγο στον εισηγητή. Παρακαλώ κύριε Βότσον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, έχω να προτείνω μια προφορική τροποποίηση στην ε, προφορική τροπολογία που συζητιέται από διάφορες πολιτικές ομάδες. Θα πρέπει να λέει προκειμένου να εφαρμόσει καθεστώτα κυρώσεων με σοβαρό τρόπο προκειμένου να αποφευχθεί η εφαρμογή διπλών ε, προδιαγραφών. Δύο μέτρων και δύο σταθμών δηλαδή. Ποιοι είναι υπέρ της προφορικής αυτής τροποποίησης, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ναι. Συμβιβαστική, μια στιγμή, όχι. Πρώτα, τροπολογία 61, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Να επαληθεύσουμε. Εντάξει, τροπολογία 61. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τώρα περνάμε στη, στην 62. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 70 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 71 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 74-75 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 76 υπέρ, κατά, μια στιγμή. Να επαληθεύσουμε εδώ παρακαλώ. Αρχίζει η ψηφοφορία για την 76 παρακαλώ. Ψηφίστε. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 77 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 78 υπέρ, κατά, αποχές θα επαληθεύσουμε για την 78 παρακαλώ. Ψηφίστε. Πέρασε τις ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. 81 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Πάλι πρέπει να επαληθεύσουμε για την 81 παρακαλώ. Ψηφίστε. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 87 υπέρ. Κατά αποχές να επαληθεύσουμε για την 87. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 88 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 89 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 90 υπέρ, κατά, αποχές, προτείνω να παληθεύσουμε για την 90. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της φοφορίας. Εγκρίνεται. 93 υπέρ, κατά, αποχές, Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά να επαληθεύσουμε καλύτερα. Ψηφίζουμε 83. 93, συγγνώμη, 93. Πέρασε τι προφορίε. Εγκρίνεται. 94 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 95 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 96 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 97 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 99 τώρα υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 100 υπέρ, κατά, αποχές να επαληθεύσουμε παρακαλώ την 100. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της φοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 11. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 12. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 107. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 108. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 109 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Αλλά να επαληθεύσουμε. 109 παρακαλώ ψηφίστε, πέρα τη φοφορίες. Εγκρίνεται. Με μεγάλη πλειοψηφία μάλιστα. Είσαστε κουρασμένοι μάλλον γιατί δεν σηκώνετε τα χέρια. 113-114 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. 115 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 117 υπέρ, κατά, μια στιγμή. Υπάρχει ένα πρόβλημα στους σοσιαλιστές μου φαίνεται. Mm γιατί ήταν αντιφατικό αυτό που ψηφίσατε. Ξανά, 117. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 13. Θέλετε για την 117. Εγκρίθηκε, εγκρίθηκε. 117. Ωραία, να επαληθεύσουμε. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Πέρα τη φοφορίες. Ορίστε, με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε. Συμβαστική 13. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 122 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 126 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 127 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 15 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 130 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 131 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 132 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 133 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 134 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται αλλά να επαληθεύσουμε καλύτερα ψηφίζουμε 134. Πέρα τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 136 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και έτσι περνάμε στην τροπολογία 5. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά αποχές να επαληθεύσουμε εδώ καλύτερα. Ψηφίστε παρακαλώ για τη 13. Πέρα της ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά. Οι σοσιαλιστές έχουν κουραστεί, μου φαίνεται. Χρειάζονται διακοπές επιγόντως. Δεν ψηφίζουν πια. Μπορείτε να μην κάνετε παρακαλώ παρατηρήσεις για τον τρόπο με τον οποίο ψηφίζουν οι σοσιαλιστές. Μα δεν ψηφίζεται, λέει Πρόεδρο. Δεν ψηφίζεται. υπέρ. Α, όχι, την κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Συμβιβαστική αριθμό 1, υπέρ. Ε. Κατά, κατά, αποχές εγκρίνεται. 19-20 τώρα, υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. 21, υπέρ κατά, αποχές. Να επαληθεύσουμε παρακαλώ. Ψηφίστε για την 21. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 22 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται νομίζω. Καλά, να επαληθεύσουμε για την 29. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα στις φοφορίες. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 34. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 35. Υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Να επαληθεύσουμε. Ψηφίστε παρακαλώ για την 35. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία αριθμός 1. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 3. Υπέρ, κατά, αποχές να επαληθεύσουμε παρακαλώ. Τροπολογία 3. Ψηφίστε. Πέρας της φοφορίας. Απορρίπτεται. τέσσερα Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και τώρα τελική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρας της Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Συγχαρητήρια κύριε Βάτσον. Τώρα θα ψηφίσουμε την έκθεση του κυρίου Σάριου Βόλσκι, εξωτερική πολιτική χώρε, Μπρικ κλπ. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. Χες εγκρίνεται. 2 συμβαστική υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Εξήντα εννέα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 80 υπέρ κατά μοχές νομίζω ότι απορρίπτεται Ογδόντα ένα, ογδόντα δύο. Ογδόντα ένα, ογδόντα δύο, υπέρ. Κατά, Όχι. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ, κατά, χες, γκρίνεται 94 υπέρ, κατά, αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται αλλά θα επαληθεύσουμε για την 94. Αρχή, τέλος. Απορρίφθηκε. 95 υπέρ. Κατά. χες Απορρίφθηκε. Όχι, εγκρίνεται, εγκρίνεται. 96 υπέρ. απαλήθευση Για την 95 ξανά. 95 ξανά. Ψήφισαν όλοι. Λείπει ένα. Λείπει ένα ή μία. Έληξε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 96 υπέρ. Κατά. Ποιες. Εγκρίνεται. 97 υπέρ. Κατά. Ποιες. Εγκρίνεται. 98 υπέρ. Κατά. Ποιες. Εγκρίνεται. 99 υπέρ. Κατά. Ποιες. Εγκρίνεται. 100 υπέρ. Κατά. Ποιες. Εγκρίνεται. 101 υπέρ. Κατά οχές εγκρίνεται 102 υπέρ κατά οχές εγκρίνεται 103 υπέρ κατά οχές εγκρίνεται συμβιβαστική 5 υπέρ κατά οχές εγκρίνεται 113 υπέρ κατά χες απορρίπτεται 114 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 6 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 116 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 117 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 7 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 126 υπέρ κατά χες εγκρίνεται συμβιβαστική 8 υπέρ κατά χες εγκρίνεται 136 υπέρ κατά χες εγκρίνεται συμβιβαστική 9 υπέρ κατά χες εγκρίνεται 145 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 10 υπέρ, κατά, εποχές εγκρίνεται. 153 υπέρ, κατά, εποχές απορρίπτεται. Επαλήθευση. Άρχισε. Έληξε. Απορρίπτεται. Εγώ έχω χρόνο, δεν με ενδιαφέρει. Άμα θέλετε να τα επελθεύσουμε όλα. 154 υπέρ. Κατά. Yes. Απορρίπτεται. 155 υπέρ, κατά, ποχές απορρίπτεται. 156 υπέρ, κατά, ποχές εγκρίνεται. 157 υπέρ, κατά, ποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 11 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 164 υπέρ, κατά, αποχές, Νομίζω ότι εγκρίθηκε, νομίζω. Τέσσερα σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, ποιες εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Πέντε υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Έξι υπέρ, κατά, Νομίζω ότι έχει εγκριθεί αλλά θα επαληθεύσουμε για την 6 ψηφοφορία. Έληξε. Απορρίφθηκε. 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. μια στιγμή ένα πρόβλημα με το ΕΛΚ για την 7 έλεγα 7 υπέρ Κατά. Αποχές. Θα επαληθεύσουμε. οι 7 ηλεκτρονικά. Έλξε. Απορρίπτεται. 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 10 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 12 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 18 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 13 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται μια στιγμή ξεχάσαμε την 11 Λοιπόν, 11 υπέρ, κατά, εποχές, απορρίπτεται. 23 υπέρ, κατά, εποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται. 24-25 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 26 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ...36 υπέρ... ...κατά... ...χες... ...εγκρίνεται... ...37 υπέρ... ...κατά... ...αποχές... ...εγκρίνεται... ...εδώ έχουμε την 38 σε δύο τμήματα... ...πρώτο τμήμα υπέρ... ...κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο υπέρ κατά εγκρίνεται. 39 υπέρ κατά χες επαλήθευση για την 39 εγκρίνεται 40 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 41-42 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται τι θέλετε να επαληθεύσουμε για το δεύτερο τμήμα ορίστε 41-42 δεύτερο τμήμα Απορρίφθηκε. 43 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 15 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 50 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ένα υπέρ, κατά, όχι, εγκρίνεται. Δύο υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η τρία καταφύπτει. Τώρα η γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης. Ανάπτ Ένα υπέρ, κατά Δεν γίνεται όλες μαζί, δεν γίνεται. Απορρίπτεται. Δύο υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. Τρία υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Τέσσερα υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Πέντε υπέρ, κατά, θα το επαληθεύσουμε αυτό, το πέντε. Το πέντε ανάπτ απορρίπτεται. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 10 υπέρ κατά χες εγκρίνεται 11 υπέρ κατά νομίζω ότι απορρίπτεται 12 υπέρ κατά χες απορρίπτεται 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 15 υπέρ. 15 είπα, υπέρ. Κατά. Ποιες εγκρίνεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Α υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Β. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. και Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. και Απορρίπτω. Τελική ψηφοφορία άρχεται ηλεκτρονικός. Ψηφίσατε όλοι και όλες. Λείπει ένα πρόσωπο ή άτομο. Έληξε εγκρίνεται πανηγυρικά. Συγχαρητήρια κύριε Σάριου Βόλσκι. Ευχαριστώ τους πάντας. Τελειώσαμε για το πρωί. Τι θέλετε κύριε Λαντσμπέργκη. Ορίστε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να κάνω μία μικρή επεξηγησούλα Γι' αυτό που με ενδιέφερε στο έγγραφο αυτό. Όταν οι χώρες BRIC παρουσιάζονται ως οντότητα, ως δύναμη, αυτό δεν ισχύει ή δεν ισχύει ακόμα. Καλύτερο θα ήταν να γίνουν διορθώσεις δεν θα γίνουν βέβαια, δεν έγιναν. Και τώρα μιλάμε για τα BRIC σαν να είναι ενιαία δύναμη. Πράγμα το οποίο είναι αναλυθές. Και δεν είναι και τόσο θετικό όπως αναφέρεται εδώ μέσα. Παραδείγματος χάρη, προσπάθησα να τροπολογήσω την το σημείο 13 ή μάλλον να υποβάλω την τροπολογία 13 όπου λέω ότι όταν επενούμε μια τέτοια οντότητα ως θετική αλλαγή ως μετακίνηση προς ένα πολυπολικό σύστημα κάτε δεν είναι αυτή η αλλαγή. Γιατί οι χώρες BRIC καταλήγουν σε μία διπολικότητα. BRIC ή οι άλλοι με επικεφαλή στην Ρωσία και την Κίνα. Πρέπει να τα αφήσουμε όλα αυτά σε μία υποσημείωση και ένα σημείο και να μην τα πενούμε τόσο πολύ αυτό το καινούργιο σύστημα. Αλλιώς θα καταλήξουμε στην περιθωριοποίησή των. Ευχαριστούμε. Τελειώσαμε για το πρωί. Θα ξαναβρεθούμε το απόγευμα. Χαίρετε.